σε συμφωνία με τις πολιτικές ομάδες προτείνω στο Κοινοβούλιο αλλαγή στην αυριανή ημερήσια διάταξη για την Πέμπτη και μάλιστα έκτακτη συζήτηση για τη θανατική ποινή στην Ινδονησία χωρίς ψήφισμα. Προστίθεται αύριο το απόγευμα ως πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Μετά τη δήλωση προβλέπεται ένας γύρος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες και η ψηφοφορία για τα κατεπήγοντα θα γίνει στις 4.30. Διαφωνείτε? Όχι. Τότε εγκρίνεται ούτως ε, τροποποιημένη ημερήσια διάταξη.